χαιρετίζω την εκλογή του κυρίου Τόκες στο Προεδρείο. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ε, ψήφου. Mr. Lambrinidis. Κύριος Λαμπρινίδης, διαδικαστικό παρακαλώ. Mr. President, just... Κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβω λίγο, τι μας λέτε τώρα, ότι για αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να μην έχει ειδική πλειοψηφία. Γιατί αν μπορείς να ψηφίσεις μόνο είτε υπέρ, είτε αποχή που να μην προσμετράτε στο συνολικό ε, αριθμό, τότε εξορισμού πάντα θα παίρνει ειδική πλειοψηφία που χρειάζεται και θα εκλέγεται ο υποψήφιος. Αυτό μας λέτε. Όπως θα θυμάστε κύριε Λαμπρινίδη, στην αρχή ε, της εκλογής του Προεδρείου είχαμε τρεις κάλπες Μάλλον, συγγνώμη, χρειάστηκαν τρει γύρι ε, ε, για να εκλεγεί ε, αντιπρόεδρος. Τότε είχαμε αυτή τη διαδικασία, σήμερα ήταν ένας μόνο υποψήφιος και επειδή πήρε πάνω από 168 ψήφους, πήρε περισσότερο από την ειδική πλειοψηφία που χρειάζεται και εξελέγει με μία και μόνη ψηφοφορία. Είναι ασυνήθιστη η διαδικασία, αλλά σύμφωνη με τον κανονισμό. Κύριε Γκέμπελς, πρώτα. Ο κύριος Γκέμπελς και μετά εσείς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να ακολουθήσατε τους κανόνες, αλλά εγώ αθρίζω. 334 υπέρ είπατε. 168 αποχές ξέρω εγώ και 287 υπέρ εγώ φτάνω σε 789 βουλευτές. Είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Άρα βία και νοθεία, όπως τις εκλογές της Γκορσική, Είναι νοθευμένη η εκλογική διαδικασία και θα πρέπει να επαναληφθεί. The explanation is, Mr. Κύριε Γκέμπερς, να σας εξηγήσω. Κύριε Γκέμπερς, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι η εξής. Παρεξήγηση έγινε. Παρανόησαν πολλοί συνάδελφοι. Ε, στην οθόνη η απόλυτη πλειοψηφία να σαν να ήταν αποτέλεσμα. Όχι. Ήταν ένδειξη. Δεν θα πρέπει να το προσθέσετε αυτό στο σύνολο των ψήφων. Η ένδειξη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ψηφοφορία. Πήρε 334 ψήφου υπέρ ο κύριο Στόκε. Είναι πάνω από εκείνο που απαιτείται και εκλέγεται. Συνεπώ. Το 168 δεν ήταν ψήφι, ούτε αποχή, ούτε τίποτα. Ήταν ε, το κατόφλι που χρειάζεται για να εκλεγεί αντιπρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη για την παρεξήγηση. Δεν ήταν σαφές τότε. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να θυμίσω μόνο ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου που προείδρευε εκείνη την ώρα μας ενημέρωσε, λέει ο κύριος Σέβεριν, ότι εκείνοι που θέλουν να ψηφίσουν αποχή και κατά έπρεπε να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό μας είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και βεβαίως αυτό μας παραπλάνησε. Πάντως, εφόσον ε, ανακοινώνεται τώρα αυτό από το Προεδρείο, είναι έγκυρο ε, και θα πρέπει να επαναληφθεί η ε, ψηφοφορία βάσει των στοιχείων και των διευκρινήσεων που μόλις μας δώσατε. was... Είμαι πεπισμένος ότι αν ξαναγινόταν η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος κατάλαβε και ψήφιζε κανονικά δεν είναι μια συνήθις ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι σαφές. Αυτό που ήταν ασαφές ήταν το 168 και που είχε μπει στην οθόνη. Αυτό σας οδήγησε σε κάποια σύγχυση. Ε, εντάξει, αν υπάρχει και άλλο θέμα, ρωτήστε τον πρόεδρο. Κυρία Σέλισιν, διαδικαστικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. ζητάμε σε σένα, E, panie Przewodniczący, no Κύριε Πρόεδρε, φοβούμαι ότι είναι όλος ανεπαρκής οι εξηγήσει τις οποίες έχετε παράσχει. Αυτό που μας δηλαδή, σχετικό με την αποχή και την ψήφο κατά, ό,τι προσμετρώνεται από κοινού. Άρα θα πρέπει να δοθεί ορισμός. Τι είπα να πει ε, η δική πλειοψηφία. Επομένως, δεν είναι ξεκάθαρο. Μέχρι να ε, δούμε τι καλύπτει ο όρος η δική πλειοψηφία, δεν είναι ξεκάθαρο το ποιο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε 387, 384 και τις αποχές. Αυτό ανακοινώθη ως αποτέλεσμα από τον πρόεδρο Μπούζεκ. Και το σύνολο, αν τα προσθέσουμε, είναι 789. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια ψήφος μετράει και ποια δεν μετράει. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Ακριβώς όπως είναι αυθαίρετο και απαράδεκτο το πώς κατανέμονται οι ψήφοι αναχώρα. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα εγκυρότητας της εκλογής. Νομίζω πρέπει να επαναληφθεί. Θα ληφθούν αυτά υπόψη, τα διαδικαστικά λέει ο πρόεδρος. Σίνκλερ, Γκέλνις, Ντέιβιτ. Παρακαλώ περιοριστείτε στο ένα λεπτό που είχε στη διάθεσή σας. Σύγκλερ. Δύο διαδικαστικά πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την εκλογή του αντιπροέδρου. Νομίζω ότι μας παρασύρατε με τις οδηγίες που δώσατε. Ε, κάποιοι θέλουν να ψηφίσουμε κατά. Δεν μας άφηνε το μηχάνημα. Άρα ζητώ επανάληψη της ψηφοφορίας και να μπορούμε να έχουμε ναι, όχι και αποχή το οποίο να εμφαίνεται κάπου. Ευχαριστώ πάντως για τη δική σας συμβολή. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν μου επιτράπει να κάνω δήλωση επί, των, επί της ε, ψηφοφορίας Για τη διαφάνεια. Ψήφισα κατά, δεν με αφήσατε να σε εξηγήσω γιατί, αλλά αυτοί που με ψήφισαν πρέπει να ξέρουν γιατί ψήφισα κατά. Παρακαλώ, θερμά να με αφήσετε να προβώ σε δήλωση σχετικά με αυτό το οποίο ψήφισα. Um, Για το πρώτο από αυτά που είπατε, Υπήρχε εδώ το προσωπικό συνεργάτη μα, ήταν εδώ και ο πρόεδρο και αν τυχόν ε, ανακύπτουν κάποιε δήματα σε σχέση με τη διαχείριση τη ψηφοφορία, αυτό θα εκπληρωθούν αρμοδίω. Δεύτερον, όσον αφορά την απλουστευμένη διαδικασία, δεν υπάρχει συζήτηση και δεν υπάρχει δήλωση επί τη ψηφοφορία. Όμω, κυρία Σινκλέρ, μπορείτε εγγράφω να προβείτε σε δήλωση επί των όσων ψηφίσετε τώρα. Έχει το λόγο, Πάρα πολύ καλά σα ε, άκουσα και πρόσεξα πάρα πολύ καλά όσα μα είπατε και είπατε ότι το 178 είναι το κατόφλι ούτω ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η ειδική πλειοψηφία αυτό μου μεταφράσανε, αυτό άκουσα, το οποίο μου φαίνεται απίστευτο. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα θεωρείται ως κατόφλι για να εκλεγεί κανείς το ίμιση αυτών που εψήφισαν ναι. Επομένως, έτσι βγαίνει η δική πλειοψηφία. 168 με 168 ψήφους έχει κανείς την ειδική πλειοψηφία. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Άρα φαντάζομαι δεν κατάλαβα καλά, δεν άκουσα καλά. Πάντως είναι παράλογη όλη αυτή η διαδικασία που έγινε. Ίσως αυτό σε άλλου είδου εκλογέ με διαφόρους υποψηφίου μπορεί να γίνει, αλλά όχι στην πλήρωση θέση θέσης αντιπρόεδρου. Το 168 λέει ο Πρόεδρο. υπολογίστηκε από τον υπολογιστή επί τη βάση αυτών οι οποίοι ψήφισαν. Και έτσι βγήκε η πλειοψηφία, επί τη βάση αυτών που ψήφισαν, των ψηφισάντων. Τι να σας πω, εγώ πήγα στο κλασικό, αλλά τι να σας πω για τα νούμερα. Uh, Ακριβώς για αυτό το θέμα. Για μια φορά, ε, πρώτη και τελευταία στη ζωή μου, ελπίζω, συμφωνώ με τον κύριο Γκόλνης. Όταν ψηφίζουν 600 ε, τόσοι, 630 βουλευτές, θα πρέπει ε, να είναι 310 τουλάχιστον. Καλά, ο συνάδελφος πήρε 334 και εξελέγει έτσι και σας παρακαλώ ε, να το διορθώσετε. Αν είναι πρόγραμμα αυτό στον υπολογιστή, σίγουρα από μαθηματικής απόψεως είναι εσφαλμένο. Ευχαριστώ. Κύριος Γκρούτε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γκρούτε. Κατά την ε, ψηφοφορία δεν μπορούσα να ψηφίσω όχι. Ε, στη δική μου τη μηχανή πρέπει να ψηφίσω ναι και μετά αποχή. Και παρακαλώ λοιπόν πώς η συσκευή μου κατέγραψε την ψήφο μου. Ε, και δεν συνέβη μόνο με μένα αυτό, συνέβη ε, και με άλλους. Δεν μπορούσε κανείς να ψηφίσει ούτε αποχή, ούτε όχι. Έπρεπε κανείς να ψηφίσει ναι. Και γι' αυτό ερωτώ. Είναι σωστό αυτό. Πολύ περιπετειώδες το σύστημα ψηφοφορίας. Παρακαλώ πολύ να επανελέγξετε πώς μετρήθηκαν οι ψήφοι. Ε, κάτι νομίζω μου οδηγεί να πιστεύω ότι αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ στο μέλλον. Καλύτερα χαρτί και κλασικά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι είχαμε 621 ψήφους και ο αντιπρόεδρος πήρε 334. Είναι η πλειοψηφία. Ας προχωρήσουμε. Και τελικά υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα που είναι επίκαιρα. Η ανεργία, ας πούμε, τώρα μην χάνουμε το χρόνο μας ε, για αυτό το θέμα. Εγώ ε, δέχομαι τις εξηγήσει σας, ε, κύριε Αντιπρόεδρε και Πρόεδρε της συζήτηση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, με πάση περιπτώσει, ας ασχοληθούμε με κάτι που είναι πραγματικά ουσιώδες. Ο κύριος Μάντερς, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω κι εγώ, η εξήγηση που μας δώσατε, που ήταν σαφής για μένα, να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη. Λυπάμαι που οι συνάδελφοι που ανεβαίνουν ε, πάντα στις ελπάξεις για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία έφυγαν τρέχοντας για φαγητό παρακαλώ να ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και να ξέρουν και εκείνοι τι γίνεται. Αυτό είναι απόφαση του Προέδρου, αλλά θα του το διαβιβάσω. Δύο ακόμα και τελειώσαμε. Η κυρία Τάιν, παρακαλώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας ε, είναι ανοιχτές και μεταδίδονται. Ε, και εδώ δώσαμε μια πολύ άσχημη εικόνα. Θα ήθελα λοιπόν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ξεκαθαριστεί η όλη υπόθεση γιατί ε, κάτι που είναι λάθος. Ε, όταν ψηφίζουν οι 600 δεν μπορεί οι 180 να είναι το όριο, ε, τουλάχιστον το ίμιση πρέπει να είναι η πλειοψηφία. Να το εξηγήσετε αυτό γραπτά στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να το κατανοήσουν και όλοι οι θεατές. Γιατί πάρα πολλοί παρακολουθούσαν σήμερα μέσω του διαδικτύου τη συνεδρίαση και πραγματικά δώσαμε μια πάρα πολύ αρνητική εικόνα. Η κυρία Ταντσίλα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, πρόεδρε, υπάρχει ένα πράγμα που δεν το κατάλαβα. Αν ήταν 334 υπέρ, τότε θα πρέπει να δείτε λιγάκι τον αριθμό των ε, αποχών. Δυστυχώς έκλεισε το μικρόφωνο της κυρίας ε, Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ε, τέλος πάντων έκλεισε αυτή η ψηφορία και πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Φτάνει. Φτάνει και εγώ θέλω να πάω για φαΐ, ο πρόεδρος. Πάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Κέλλη. Ε, πρώτος ο κύριος Γκάλαχα. Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ, αλλά δεν εξεπλάγει από την ε, συντριπτική υπερψήφιση αυτής της ε, έκθεσης. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σημαντικά από το μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση του Λονδίνου για να προαχθεί η κοινωνική ανάπτυξη και στις ε, δύο πλευρές των ε, συνόρων. Πρόκειται λοιπόν για μια επένδυση ε, της τάξης πάνω από 2 δις ευρώ αν λάβουμε υπόψη μας ε, και τον πολλαπλασιαστή. Εγώ ο ίδιος είμαι από μια παραμεθόρια περιοχή και ως εκ τούτου γνωρίζω πολύ καλά το ρόλο που είχε αυτό το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής διαδικασίας. Πολλές ε, θέσεις εργασίας ε, συστήθηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου και επίσης ε, δημιουργήθηκαν και ευκαιρίες απασχόλησης σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές. Εγώ κύριε Αντιπρόεδρε πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το αποτελεσματικό πρόγραμμα. Επόμενος η επόμενη, η κυρία Μπουμπά Μπαρμπάμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την ε, πρωτοβουλία αυτή γιατί βασικό στόχος είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει τη συμφιλίωση και την ειρήνη ε, στη Βόρεια Ιρλανδία και στις παραμεθόριες περιοχές για να μπορέσει κανείς να χτίσει τη συμφιλίωση και ε, την επικοινωνία μεταξύ αντιτιθυμένων κοινοτήτων και λαών. Στη χώρα του Βάσκο Νεοσκάδη ακόμα ε, υφιστάμεθα τη βία τη τρομοκρατία και ελπίζω η ΕΤΑ να έχει καταλάβει και να ακούει τη φωνή των Βάσκων που έχουν κουραστεί και τους δουν να εγκαταλείψουν τα όπλα. Περιμένουμε μια οριστική ε, κατάπαυση του πυρός και παράδοση των όπλων να εξαγγείλουν για να οικοδομήσουμε και στη χώρα των Βάσκων ειρήνη και συμφιλίωση που τόσο πολύ λαχταρούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καμιά χώρα δεν έχει πληγεί τόσο πολύ όσο η Ιρλανδία από αυτές τις εξαιρέσεις. Ο Πρωθυπουργό αποφάσισε όσο πιο σωστά γινόταν. Και όλοι, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έσφιξαν το ζωνάρι ακόμα και ακόμα και άνεργοι. Τώρα μας λένε για περισσότερες περικοπές και λένε να κάνουν και οι Έλληνες το ίδιο, να γίνει εξαίρεση για τους Έλληνες και επίσης τώρα θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε ε, να σωθεί η Ελλάδα και καταλήγουμε να πληρώνουμε ακόμα περισσότερο από τα άλλα μέρη της Ευρωζώνης για την Ελλάδα και οποιοδήποτε οικονομολόγος θα έλεγε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδου περιθώριο στην Ευρωζώνη, να γίνει κάποια υποτίμηση και έτσι να αποκατασταθεί η κατάσταση και να μην καταδικάζουμε τους λαούς της Νότιας Ευρώπης σε φτώχεια, σε, σε, σε, λιτότητα και απ' την άλλη να πρέπει να βάλουμε βαθιά στο τσέπη αυτοί που είναι στην Βόρεια Ευρώπη. Thank you very much. Nicholson. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα να προβάσω επεξήγηση ψήφου, όμως άκουσα τον κύριο Πέσλε, τον κύριο Άνταμς, υποσυγητής, και είπε για τις συμβολίες στην ειρήνη Ευζωρία Πρόεδρε, ο κύριος Άνταμς και ο δόκτωρος Πέσλε φέρανε πολλά, αλλά όχι και την ειρήνευση. Ο Τζον Χιούμ μίλησε για το πώς μπορεί να έρθει η ειρήνη. Εγώ πάντως υπερψήφισα την έκθεση γιατί θεωρώ ότι σήμερα στην Βορειοελλανδία χρειαζόμαστε ακόμα στήριξη για να παγιώσουμε αυτά που πετύχαμε. Δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο ότι υπάρχει θα διατηρηθεί η ειρήνη. Πρέπει να το δουν και οι δύο πλευρές Κοίτατε τι έγινε πρόσφατα από αυτούς που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν και πάλι την κατάσταση. Κούσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν από τους 334 ευρωβουλευτές που υποστήριξαν τον κύριο Λάσλο Τόκερς ε, για την εκλογή του ως αντιπρόεδρος. Όταν ήμουν νέος, ήμουν στην Αλληλεγγύη το 1989, στην Πολωνία, δημοσιογράφος και έγραφα για τις σφαίρες της Εκουριτάτη του Τσαουσέσκου στις οποίες κατέπνιξαν στο αίμα ε, την επανάσταση στη Ρουμανία. Το είπε και ο Λάσο το Δεκέμβριο του 89 στην Τιμισόαρα. Και πραγματικά με θλίβει και με πονάει και μένα αυτό που έγινε σήμερα. Τα σφάλματα στη ψηφοφορία που οδήγησαν σε γενική αντιπαράθεση. Ε, αν κάποιος ε, αμφισβητήσει την εγκυρότητα αυτής της ψηφοφορίας, ας επαναληφθεί. Είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για το συγκεκριμένο άνθρωπο και μάλιστα θα πάρει ακόμα περισσότερες ψήφους. Θα έχει ακόμα καλύτερη ψηφοφορία και κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την αξία και ε, το πρόσωπο του κυρίου Τόκες. Ο πρόεδρος, θέλω να κάνω και εγώ μερικά σχόλια. Εγώ ήμουν ανέκαθεν ε, υποστηρικτής και θαυμαστής του Πάστορα Τόκες, ε, του επισημωτά του, ε, και κατά τη διάρκεια ε, της δικτατορίας του Τσαουσέσκου και λυπάμαι που έγιναν αυτά τα επεισόδια. Εξελέγει όμως κανονικά ο άνθρωπος και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, πάμε τώρα στην έκθεση Μαρινέσκου. Έχω μία επεξήγηση. Ο κύριος Αντωνιώτση. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ στήριξα την έκθεση Μαρινέσκου και δράτω με τις ευκαιρίες για να τον ευχαριστήσω γιατί θεωρώ ότι η σωστή μεταφορά των εμπορευμάτων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα αλλά ακόμα και για την επιβίωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να στηρίξουμε ε, την βούληση του εισηγητή να επαναφέρει κάποιες ε, παραγράφους οι οποίες μπορούν και να εγκριθούν σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έκθεση Μάρτιν, ο κύριος Χάνον. Πρόεδρε, όταν ξεκινήσαμε σήμερα την ψηφοφορία, αντιμετωπίσαμε μια διαδικασία που ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Κατεγράφονται μόνο οι θετικές ψήφοι. Ε, τελικά όμως ε, αυτή την προσέγγιση έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, διάφορα δημοψηφίσματα. Συνεχώς απορρίπτεται το το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα ε, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και κάθε φορά η αντίδραση ήταν να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίσει παντελώς ε, τις αντιρρήσεις των πολιτών και να ακούει μόνο ε, το ναι. Τώρα λοιπόν ε, τι βλέπουμε αυτή τη διαδικασία, την ε, έχουμε θεσμοθετήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν κάποιος διαφωνεί αυτό δεν μπορεί να ε, καταγραφεί. Και διερωτάμε, άλλα, εσείς τι είδους όχι κατανοείτε. Καμάλ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχουμε αυτή την έκθεση που αφορά την ε, προσαρμογή της διαδικασίας ε, της δικής μας και του κανονισμού στη Συνήθεια Λισαβόνας. Οι περισσότεροι νομίζω από εμά δεν ξέρουν τη λέει της Λισαβόνα κάτι το οποίο φυσικά και έχει σημασία στην καθημερινή ζωή. Ε, για, τον κόσμο. Κοιτάξτε, είδατε τι έγινε για τη Σωτήρια της Ελλάδας, είδατε τι, τι συζητήθηκε για το άρθρο 122 της Συνήθισης Λισαβόνα στο Συμβούλιο. Υποτίθεται ότι αυτό το άρθρο εκφράζει την αλληλεγγύη. Ε, αλληλεγγύη προς μία χώρα όταν έχει κάποια δυσκολία για κάποιο προϊόν, για, κάποια, για, την, για κάποιο ενεργειακό θέμα ή όταν πλήσεται από κάποια θεομηνία. Δεν είναι δυνατόν να επικαλεστεί κανείς αυτό το άρθρο ως δικαιολογία για κάποιο κράτος μέλος, μέλος Ευρωζώνης ή όχι, ούτως ώστε να σωθεί κάποια χώρα η οποία όμως μόνη της προκάλεσε τα δεινά της και ε, δεν είναι κάτι το οποίο έχει υποστεί λόγω ειδικών ε, συνθήκων και περιστάσεων. Άρα θα πρέπει να ξεθαριστεί τη λεσνίκη της Λισαβόνας και να μην ε, ξεπαραδιαζόμαστε για να αφορούμε αυτούς οι οποίοι πέσαν στον εαυτό τους τα οικονομικά δυνάτους. Ο επόμενος. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την του κανονισμού. Πάντοτε το θέμα είναι το πώς θα, θα περισταλούν τα δικαιώματα των, των, των, των των μειονοτήτων, των, των μη προνομιούχων, ημών ε, δηλαδή. Ποιο ένα χρόνο που τα συζητάμε σε σχέση με το άρθρο 24. Τι γίνεται με τους μη εγγεγραμμένους, τους ανεξαρτήτους. Ε, διότι... Ε, συγγνώμη, αλλά άκουσα αυτό το οποίο είπατε ότι δεν είναι δυνατόν. Είναι από τα πιο ανόητα πράγματα που έχω ακούσει κατά την κοινοβουλευτική μου βία, ότι δεν είναι δυνατόν να, να γίνει έτσι. Ε, εγώ είμαι μια εγγεγραμμένο επειδή το ζητώ και εσεί όμω και εσεί μια εγγεγραμμένο γιατί δεν σα υποστηρίζει κανένα. Σα προ, προδώσαν οι συνεργάτε του κόμματό σα. αυτό, αυτό πάνω από δημοκρατία. Θα πρέπει αυτοί που ε, να ορίζονται έτσι οι εκπρόσωποι των μη εγγεγραμμένων. είναι κοροϊδία για άλλη μια φορά. Ο κύριο Μάρτιν κάθισε και το σκέφτηκε αυτό με του εκπροσώπου των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων. Γιατί δεν κάθισε να σκεφτεί για τον προηγούμενο, προηγούμενο κανονισμό, την ανθεώρηση του κύριο Κόρμπετ, ο οποίο τώρα ο κύριο Κόρμπετ έφυγε αλλά γαλλικά και ο οποίο μαυρώθηκε, έφαγε μαύρο και δεν εξελέγει στι εκλογέ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι η δική σα ε, εκδοχή για μη γραμμές, δεν ισχύει. Ο κύριος Κλάι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 86 της έκθεσης ε, Μάρτιν ορίζει ότι ο εκπρόσωπος των μη στη διάσκεψη των Προέδρων δεν εκλέγεται από τους ίδιους τους μη εγγεγραμμένους, αλλά ορίζεται, λέει, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για ποιο λόγο, γιατί υποτίθεται ότι δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ των μη εγγεγραμμένων μελών. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ερωτώ. Στο Κοινοβούλιο, εδώ, που εκλέγεται ο πρόεδρος ε, δεν είναι και αυτό συνενετικός, γι' αυτό έχουμε εκλογή με τρόπο δημοκρατικό. Και ο εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να εκλέγεται. Και τώρα ερχόμαστε σε μια κατάσταση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίθεται ότι είναι κοινοβούλιο Μίκη Μάους, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος ορίζει ένα εκπρόσωπο των αντιπάλων του ε, και μάλιστα αν είναι αντιπροσωπευτικός και όχι. Και ρωτώ με ποια βάση, πού είναι αντιπροσωπευτικότητα. Τι είναι, άμα τον αγαπάει, είναι φίλος του, έχει προσωπική συμπάθεια για τον Α ή τον Β μη εγγραμμένο. Με ποια κριτήρια θα ορίζει ο πρόεδρος την εκπροσώπηση των μη εγγραμμένων στη διάσκεψη των πρόεδρων. Θα ήθελα παρακαλώ να μου ε, κάνει δήλωση ο πρόεδρος πριν την ψηφοφορία, αλλά φυσικά δεν μας δώσατε αυτό το δικαίωμα. Λυπάμαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάστορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε το πώς θα προσαρμοστεί ο κανονισμός μας στην Εκκλησία της Λισαβόνας τι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν, αλλά είπαμε και κάποια κενά που υπάρχουν στη διαδικασία. Κάποια κενά τα οποία μα οδηγούν σε τέτοια παράδοξα αποτελέσματα όπω έγινε σήμερα και δεν καταλαβαίνω. Ο κάθε ένα αντιπρόεδρο αλλιώ τα είπε. Ο κάθε ένα προεδρεύων μάλλον αλλιώ τα εξήγησε. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι δεν έγινε σωστή καταμέτρηση τη ψήφου του. Άρα θα πρέπει να το ξανακάνουμε στην πληροφορία. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, ξέρετε, δεν μπόρεσαν καν να επαληθεύσουν κατά πόσον έγινε σωστή καταμέτρηση αυτού που ψήφισαν. Και ο κύριος Τούρκης επίσης. Και ο Στόκιος επίσης ε, ε, θα ενδιαφέρονται. Είναι προς το συμφέρον του να ξαναγίνει ε, αυτή η και να διασκεδαστεί κάθε εμβολία. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε μετάσταση του καρκίνου, του ελληνικού. Πάει τώρα και αλλού στη Μεσόγειο. Τώρα λένε για σωτηρία της ισπανικής οικονομίας. Τι λέει, κάνει ο κ. Φανρομπάιτ, τι έγινε με αυτά τα 750 εκατομμύρια τα οποία είπαμε ότι θα πάνε στο Ταμείο για Σωτηρία Οικονομιών, δεν θα φτάσουν. Αντί για εγχείρηση, και αποκοπή του άρρωστου μέλους διαλέξαν τη χημειοθεραπεία. Το αποτέλεσμα αδόκιμο, αβέβαιο. Τι θα γίνει με την οικονομική διακυβέρνηση, τι θα γίνει με, την, ε, με αυτό το οποίο πρότεινε ο κ. Φανερομπάη. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι φόρε στις συναλλαγές, ε, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα κόλπα, ούτω ώστε να είναι δυνατόν να υπάρξει ρευστότητα και να συνεχιστεί η επιβίωση των οικονομιών και καθόλου τον τρόπο να υπάρχει ε, κάποιο, κάποια μέθοδος να, γίνει κάποια η υποτίμηση και να ανορθωθούν οι οικονομίες. Όλα αυτά όμως είναι μια μεγάλη θυσία για να σωθούν κάποιοι οι οποίοι μετήλθουν αθέμητα μέσα. Έκθεση Κάσμαν λέει ο πρόεδρος. Μαστέλα. in occasione del vertice del millennio del 2000 οι πιο πλούσιες και οι πιο φτωχές χώρες ε, στη διάσκεψη κορυφής ε, είπαν ότι θέλουν μέχρι το 2015 να υλοποιηθούν κάποιοι στόχοι, να περιοριστεί η πείνα, να προστατευτεί το περιβάλλον, να ενισχυθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς πιστεύουμε ότι τώρα πλέον η Ευρώπη είναι ένας ε, σημαντικός παίκτη και εκείνη καλύτερα να αναλάβει ένα καθοδηγητικό ρόλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβονία ότι τα τελευταία χρόνια ε, πράγματι βοηθήσαμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, όμως ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η διεθνής κρίση αναγκάζει ε, πάρα πολλές αναπτυγμένες χώρες να περίσουν τους προβλησμούς τους για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες. Και θεωρώ κύριε Πρόεδρε, εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρξουν καινοτόμοι μηχανισμοί, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν την πολιτική για να υλοποιηθούν οι στόχοι που είναι ανάπτυξη, αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και ε, δικαίωμα στην ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, αυτό κατά την άποψή μας είναι η σημαντικότερη πρόκληση. Grazie Presidente. Εγώ κύριε Πρόεδρε υπερψήφισα την έκθεση Κάσμαν γιατί θεωρώ ότι είναι ευθύνη αυτού του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμών να σεβαστούν τις υποχρεώσεις απέναντι στα άτομα τα οποία βρίσκονται κυρίως στην Αφρική. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 2015 και να μην ε, ξέρουμε ότι έχουν επιτευχθεί οι οκτώ μας στόχοι. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας δεν πρέπει να ξεχνάμε υπάρχουν δισεκατομμύρια άτομα που υποφέρουν και που δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα ε, στην ανάπτυξη. Η διαγραφή του δημόσιου χρέους, ε, ενίσχυση ε, των προσπαθειών για καλή διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης το οποίο κατά την άποψή μα δεν πρέπει να αναπληθεί περαιτέρω γιατί αλλιώς θα υπάρξουν και άλλα ανθρώπινα θύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ε, διερμηνείς. Αναβολή μέχρι, διακόπτη συνεδρίες μέχρι τις 3.